που ο απασχολούμενος έχει, λαμβάνει οδηγίες σε καθημερινή βάση και ε, αυτό γίνεται στην χώρα που δουλεύει και όχι εκεί όπου ε, είναι η, ε, ο εργοδότης. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνει η συζήτηση. Στην έκθεση Φράγα Στέβες και δίνω το λόγο στην κυρία Φράγα Στέβες. I'm sorry to Mr. Mato. Ο κύριο Μάτο έχει το λόγο. Μιλώ εξ ονόματος ε, της κυρίας Φράγα που δεν μπόρεσε να ε, παρευρεθεί. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα ε, της αλληλευτικής πολιτικής στην περιοχή Ειρηνικού μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτικής αλίας, όπου θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας αν θέλουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα για την περιοχή του Ειρηνικού και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια ενδιάμεση ε, συμφωνία με την Παππού Νέα Γουινέα και αφορά και όλες τις ε, περιοχές ε, του, της, περιοχ, χώρες της περιοχής αυτής. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο το 2% της ε, πολιτικής της αναπτυξιακής κινείται προς αυτή την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι πόροι στον ειρηνικό και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το 2011 στον κεντρικό και δυτικό ειρηνικό υπήρξε μεγαλύτερη ε, ποσοστή αναλογία που αφορά την, ε, το αλίευμα τα αλλιεύματα αυτά και το Μπανουάτου και τα Φίτζι βρίσκονται ε, στην λίστα των χωρών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί αυτές οι αποφάσεις. Ο αλλιευτικός ε, στόλος είναι πολύ χαμηλός και γι' αυτό πιστεύουμε ότι για τα τονοειδή έχει μειωθεί η παραγωγή. Χωρίς να ξεχνάμε ότι με το Κυριμπάτι έχει συναυθεί διμερής ε, συμφωνία και με τις νήσους του Σολομόντα έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει η συμφωνία και γι' αυτό ε, ήρθαμε σε επαφή και με τις νήσους Κουκ διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αλευτικός μας στόλος κινείται και σε αυτή την περιοχή και πολύ κοντά στη Λατινική Αμερική. Η αλληλεία είναι ένας από τους λίγους τομείς που, έχει, που είναι ύψης της σημασίας για αυτές τις χώρες και η ενδιάμεση συμφωνία επετεύχθη και για τα μεταποιημένα και ημιμεταποιημένα προϊόντα, όπου υπήρξε μια εξαίρεση. Και εκεί υπήρξαν ειδικέ συμφωνίε για το δασμολογικό καθεστώς. Μιλάμε λοιπόν για συνολική εξαίρεση ως προ τα νοπά και τα κατεψυγμένα προϊόντα. Μιλάμε για μια στρατηγική μέσο και μακροπρόθεσμη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, νέες ε, συμφωνίες με τις νήσους Κου και του Βαλού και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον νησιωτικό χαρακτήρα αυτών των περιοχών και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να, ε, δεχτούμε, να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλία, όπως ήδη έχει οριστεί. Μέσο και μακροπρόθεσμα θα πρέπει η Επιτροπή να ορίσει μια περιφερειακή πολιτική με μια συμφωνία που θα ορίσει τους όρους πρόσβασης του αλλιευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας στον τομέα της αλίας και επίσης μία ε, διαχειριστική τακτική έτσι ώστε να μην υπάρξει παράνομη αλίευση ιδιαίτερα σε σχέση με τις περιοχές αυτές. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα που να εγγυηθούν την διαφάνεια και τον συμπληρωματικό χαρακτήρα της αλίας αυτής. Θα πρέπει να εξεύρουμε τρόπους για να δοθεί και να βρεθεί ένας ε, διάβλος για τα μέσα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και συμφωνίες που να προωθούν τα συμφέροντα της περιοχής. Επίσης, χρειάζεται ένα απότερο στάδιο ανάπτυξης καθαρά περιφερειακής μέσα στα πλαίσια μιας ε, πολυεθνικής συμφωνίας για την μελλοντική συμφωνία για την πρόσβαση της κοινοτικής αλίας στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I give the floor to Mrs. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η Επίτροπος Δαμανάκη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Φράγκα και την Επιτροπή Αλίες για τη σημαντική αυτή έκθεση καθώς επίσης και τον ε, συνάδελφο ο οποίος παρουσίασε την έκθεση αυτή. Ξέρετε ότι στην περιοχή του κεντρικού και δυτικού ειρηνικού υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά αποθέματα τόνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικότατος εισαγωγέας ηχθείων προφανώς έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα αλλιευτικά στην περιοχή αυτή. Να σε επενθυμίσω τις σημαντικές προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή δράση στον ειρηνικό πρώτον. Βιώσιμη αλία, βάσει επιστημονικών δεδομένων, δεύτερον καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας και τρίτον δημιουργία και βελτίωση των ελευτικών ικανοτήτων των μικρών ισιωτικών κρατών. Σε σχέση με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξωτερική διάσταση τη κοινή ελευτική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει την, προώθηση, τη βιώσιμη, υπεύθυνη και διαφανού αλίας στα ύδατα των τρίτων, των τρίτων χωρών. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε την ε, εφαρμογή περιφερειακών στρατηγικών για τη βιώσιμη αλία στον ειρηνικών. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τις ε, βασικές αυτές αρχές και τους ίδιους αυτούς βασικούς στόχους σε αυτή την περιοχή. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή αγορά εξηγεί πραγματικά και την έντονη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κεντρική και στον κεντρικό και δυτικό ειρηνικό, καθώ επίση και στα σχετικά περιφερειακά συμβούλια, μολονότι η συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλή. Όπω λέει και η έκθεση αυτή, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Ως προς αυτό λοιπόν ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τα συμπεράσματα του νέου πρωτοκόλου για την σύμπραξη αλληλευτικής συμφωνίας με το Κυριμπάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της αρχής μπορεί να αποδεχθεί τα όσα περιλαμβάνονται στην Συμφωνία Ναούρου, αρκεί αυτή να εφαρμοστεί βάσει συγκεκριμένων προποθέσεων, οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Θα πρέπει οι διατάξεις αυτές να είναι διαφανείς και θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν προκειμένου πραγματικά να ανταποκριθεί στους στόχους του και θα πρέπει να συνάδουν απόλυτα με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται τόσο στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες όσο και στην ανοιχτή θάλασσα. Η Αλία διαδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για κάποια μικρά νησιωτικά κράτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις δικαιολογημένες φιλοδοξίες των κρατών αυτών, αρκεί όμως να σέβονται τους βασικούς στόχους της βιώσιμης αλίας και της χρηστής διακυβέρνησης. Όπως λέγεται και στην εκθεσή σας, οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην περιοχή έχοντας μία συνοχή ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ακριβώς να προωθήσει αυτή τη συνοχή στις πολιτικές της, προκειμένου να καταφέρουν να ενσωματωθούν καλύτερα οι πολιτικές αλίας με τις πολιτικές εμπορίου, καθώς επίσης και αναπτυξιακής βοήθειας στις περιοχές αυτές. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να χαιρετήσω για άλλη μια φορά την πολύ καλή αυτή πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Δαμανάκη. Ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημέρα διάταξη είναι η έκθεση Σαλαβράκου περιορισμή στην Αλία και στα χωρικά ύδατα Μεσογείου και